Έχουμε το θέμα των επεξηγήσεων ψήφων στην ημερήσια διάταξη. Ας τις κάνουμε τώρα. Ο κύριος Πόσπισιλ ζήρη. Ε, απουσιάζει ο κύριος Πόσπισιλ. Η κυρία Παλώμα Λόπες Μπερμέχο. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο Γιούνκερ. Όπως εμφανίστηκε σε ένα πρόεδρος κάποια πολιτική επιτροπή, Οπότε αυτό το οποίο χρειάζεται είναι, ναι, να ε, παρουσιάζεστε έτσι και με να έχετε τη μάσκα του τεχνόκρατα και είπατε ότι θα υπάρχει μεταρρύθμιση για το ευρώ, θα υπάρχει κάποια απελευθέρωση. Ο δρόμος που θέλετε ουσιαστικά είναι να περικόψετε τα δικαιώματα των εργαζομένων ή να τα στερήσετε περιεχομένου. Και οπότε θα πρέπει να μας εξηγήσει κάποιος που είναι η καινοτομία των προτάσεων. Το, το, η μόνη καινοτομία είναι ε, ο ελάχιστος μισθός, όπως είπα, τα καθήκοντα τα καθήκοντά του. Οπότε θα πρέπει να δούμε πού θα βρούμε τους πόρους, γιατί είπαμε πέσαν οι μάσκες στην υπόθεση της Ελλάδος. Οπότε ο κυρίαρχος ε, νόμος είναι η αγορά και υπήκουν σε αυτόν όλοι οι λαοί. Να του να πει Γιούνκερ. Ε, εγώ δεν θα τον αφήσω να προχωρήσει με τη δική μου ψήφο και την ψήφο της αριστεράς. Μπάλτσο. Πρόεδρε. Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής. Δεν μπόρεσα να το υπερψηφίσω. Το καταψήφισα αναγκαστικά. Καθώς το ψήφισμα δεν δίνει ενδείξεις για το πώς σκοπεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανταπόκριση της ε, στην ε, οικονομική κρίση περιορίζεται στην κεντρική διαχείριση. Αφαιρεί από τις εθνικές κυβερνήσεις και τα εθνικά κοινοβούλια τη δυνατότητα να αποκαταστήσουν τις δημοσιονομικές ισορροπίες και δεν δίνει ελπίδα στα κράτη-μέλη της περιφέρειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχο δεν έχει να λύσει το μεταναστευτικό, αλλά μόνο να θεραπεύσει τα συμπτώματά του. Υποστηρίζεται απερίφραστα την συμφωνία εμπορικών σχέσεων και επενδύσεων με τι ΗΠΑ. Μια και είχα μόνο ένα λεπτό, θα σταματήσω. Ήταν απαράδεκτο πάντω το ψήφισμα. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μαμίκινς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ευρωπαϊκή οικονομία δεν αναπτύσσεται, διότι έχουμε ύφεση. Η ύφεση με χαμηλή ζήτηση, χαμηλό επίπεδο επενδύσεων, Πώς μπορούμε να ελπίζουμε σε ανάκαμψη της ζήτησης εφόσον υπάρχει τόσο υψηλή ανηλικία σε τόσα κάτι μέλη, ιδίως μεταξύ των νέων. Αυτοί που δεν έχουν δουλειά δεν έχουν και αγοραστική δύναμη. Πολλοί έχουν τεράστια δάνεια και πρέπει να δώσουν μεγάλο μέρος του εισοδήματό τους στις τράπεζες. Γιατί εισόδημα τελικώς μιλάμε. Ε, χιλιάδες επί χιλιάδων Ευρωπαίοι εργάζονται αλλά δεν κερδίζουν αρκετά. και η ε, μόνη τους μέρημνα είναι μήπως απολυθούν. Δεν μπορούν να εξοικονομήσουν χρήματα. Ε, γι' αυτό είναι πολλοί τομεί όπου περικόπτονται θέσει εργασία, δεν υπάρχει σταθερότητα και είναι σημαντικό στο πρόγραμμα εργασιών τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στηρίξει τη δημιουργία θέσεων απασχόληση και τη συμπερίληψη στην αγορά εργασία. Αυτό είναι ο μόνο τρόπο να ξεφύγουμε από την κρίση και την ε, ύφεση. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ τοποθετήθηκα υπέρ του προγράμματο εργασία Ευρωπαϊκή για το 2016 γιατί κατά τη γνώμη μου την ταπεινή αντιστοιχεί σε όλε τι λύσει που αναζητούμε για το περιβάλλον, την οικονομία κλπ. Επίση, ε, θεώρησαμε πάρα πολύ θετικό το ότι κατανόησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποιε είναι οι ευθύνε τη. Και κυρίω ε, όσον αφορά αυτή την ανθρωπιστική κρίση. Εγώ να αναφανδόν υπέρ. Οπότε και ακριβώ επιψήφισα το πρόγραμμά τη, διότι είναι ε, ε, αυτό το οποίο περιμένουμε και για τους περιβαλλοντικούς πρόσφυγες όπως τους λέμε, γιατί έχει πληγεί από και ξηρασία η χώρα τους. Και οπότε είμαι υπέρ και ελπίζω ότι όλα αυτά το πιάνει ανακοινώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα τα ε, τηρήσει και οπότε θα μπορέσει να μας ετοιμάσει να μηνθούμε κατά τις επόμενες κρίσεις ο Πρόεδρος. Σας ενημερώνω ότι έχω